Okay, colleagues, I'll get started. I know we're a bit thin on the ground, but I will get started anyway. Call the meeting to... Ξεκινάμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε την ημερήσια διαταξή. Αν συμφωνείτε, μπορούμε να περάσουμε και στο επόμενο σημείο, έγκριση πρακτικών 26-27 Νοέμβρη και 3 Δεκέμβρη. Συμφωνούμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο 4. Απλοποίηση της μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων ταξινομημένων σε άλλο κράτος εντός της ενιαίας αγοράς επί της ουσίας ΣΥΜΚΟ. Και η συγκεκριτής μας είναι ο κ. Σπίρκερ. Ο κ. Σπίρκερ. Um- Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, συζητάμε για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών σε σχέση με την απλοποίηση μεταφορά των μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλη χώρα μέλο εντό ενιαία αγορά. Θα ήθελα λοιπόν να σα πω ευθύ εξ αρχή ότι δεν υπάρχουν κάποια περίπλοκα θέματα εδώ. Κυρίω έχουμε τέσσερι στόχου ω νομοθετική προσπάθεια. Να διασφαλίσουμε δηλαδή την ελεύθερη μεταφορά των οχημάτων σε όλη την ενιαία αγορά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω θα ωφελήσει όλους αυτούς που εποφελούνται της κινητικότητας και είναι ένα θετικό μήνυμα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει προς τα έξω. Δεύτερος στόχος που είχαμε είναι το να μειώσουμε το διοικητικό βάρος και αυτό βεβαίως θα οδηγήσει σε μια εξοικονόμηση διοικητικού κόστους 1,5 περίπου δις ευρώ Τρίτος στόχος που είχαμε είναι το να διασφαλίσουμε την οδική ασφάλεια επειδή οι προδιαγραφές όλες τις χώρες μέλη θα εναρμονιστούν περίπου στο ίδιο επίπεδο. Και τέταρτος στόχος είναι μέσω της ανταλλαγής δεδομένων να χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία ώστε να καταπολεμήσουμε τις αυθαιρεσίες και την κλοπή γράφων ταξινόμησης. Γενικά λοιπόν ήταν μια αξιόλογη θα έλεγα πρωτοβουλία με κάποιες προτάσεις που έχει καταθέσει η Κομισιόν βεβαίως και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Σκιώδη, τους Σκιώδης. Είχαμε δύο έντονες και γεμάτες συναντήσεις όπου ανταλλάξαμε απόψεις και όπου χρειάστηκε να έρθουμε σε συμβιβασμούς. Κάποιοι αφορούσαν το χρονικό πλαίσιο και είχαμε και κάποιε απαραίτητε διευκρινήσει λόγω των διαφόρων κανόνων που ισχύουν στι διαφορέ χώρε μέλη. Βεβαίω. τώρα δεν θέλω να επισταθώ σε λεπτομέρειε για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά τέλο πάντων τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων με τους κοιόδης εισηγητής οδήγησε στο να κατατεθούν τελικά λίγε τροπολογίες και που εστιάζουν κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Και νομίζω ότι Όλοι συμφωνούμε ότι αυτό είναι θετικό. Είχαμε μόνο 33 τροπολογίες και από αυτές τις 33 τροπολογίες τελικά κάποιες από αυτές αποσύρθηκαν κιόλα. Επειδή κάποια από τα θέματα που κάλυπταν οι τροπολογίες βρισκόταν ούτως ή άλλως στην έκθεση ή τέλος πάντων περιλαμβάνονταν στην αρχική πρόταση της Κομισιόν. Οπότε δεν υπήρχε ανάγκη να προληφθούν στι τροπολογίε αυτά τα σημεία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω αυτού του συναδέλφου που το κατανόησαν αυτό και απέσυραν τι τροπολογίε του. Είχαμε κάποιε τροπολογίε οι οποίε κατατέθηκαν και οι οποίε μα βοήθησαν να διευκρινίσουμε κάποια θέματα ορολογία. Βεβαίω αυτέ θα περιληφθούν, το συμφωνήσαμε αυτό. Και υπήρξαν και λίγε τροπολογίε οι οποίε που συμφώνησαν και οι σκιώδεις να απορριφθούν επειδή θεωρήσαμε ότι αυτές οι τροπολογίες δεν θα ήταν εφαρμοστές ή εφικτές να εφαρμοστούν. Οπότε θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε για επαλήθευση κατά πόσο ποια μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν και αν χρειαστεί θα πρέπει να λάβουμε περαιτέρω μέτρα συμπληρωματικά. Νομίζω ότι όλοι συμφώνησαμε αυτή τη γενική αρχή και γι' αυτό ακριβώ το λόγο στην έκθεσή μα έχουμε πάρα πολύ λίγε τροπολογίε οι οποίε τελικά έτυχαν αποδοχή. Και πάρα πολύ λίγε τελικά που νομίζω θα πρέπει να απορρίψουμε και οι σκιώδεις ε, αποδέχτηκαν επίσης και το αιτιολογικό μια αποδοχή ή απόρριψη και αυτών των τροπολογιών. Του ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ευχαριστώ και του διάφορου ε, συμβούλου μα και εμπειρογνώμονε που μα υποστήριξαν στην δουλειά μα. Αυτά ήθελα να σα πω εγώ και προσλέπω βεβαίω ε, ερωτήσει και στη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λέει ο πρώτο, κ. Ντιμπάκα. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια των δύο ε, συναντήσεων του τους Έχω υποβάλει εγώ δύο ε, σημαντικές κατά τη γνώμη μου τροπολογίε. Μία ε, όπου τονίζεται ότι κατά κάτι μέλη θα πρέπει να επιβλέπουν τις αρχές ταξινόμησης και ότι αυτές λειτουργούν όπως πρέπει. Σε ό,τι αφορά και την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφουν και αυτή σημαντική. Μετά, ε, σε ό,τι αφορά την μεταφορά σε άλλο κράτο μέλο, θα πρέπει να γίνεται εντό τριών μηνών. Η Επιτροπή είχε προτείνει του έξι μήνε. Θεωρούμε ότι είναι ε, υπερβολικό το, χρονοδιάγραμμα. Ε, φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό θα ακολουθήσουμε τον εισηγητή. Νομίζω ότι η προσπάθεια του ήταν πολύ καλή και εργάστηκε πολύ καλά με σωστή προσέγγιση για να ε, επικεντρωθεί στα ζητήματα που αφορούν ε, στις μεταφορές ε, και επικεντρώθηκε ιδιαίτερα και στην προστασία δεδομένων που για την ομάδα μου είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Ε, χωρίς να ξεχνά και την, την ανάγκη απλούστευσης των διδικασιών για τον καταναλωτή. Και θεωρούμε ότι θα είναι πολύ εύκολη η ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Μπραντμπορν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Βέρκερ. Ε, πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ βεβαίω ότι αυτό προκύπτει από μια έκθεση που είχε παρουσιάσει η Επιτροπή Εσωτερική Αγοράς για τα 20 μεγαλύτερα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Και σίγουρα είναι κάτι θετικό το ότι προσπαθούμε να δισκεδάσουμε ε, αυτές τις ανησυχίες. Επομένω, ε, και στηρίζω αυτή την προσπάθεια δεν θα ήθελα να καταλήξουμε σε υπερβολικό γραφειοκρατικό φόρτο ε, που θα βαρύνει τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Ε, ήδη είναι πολύ υψηλό το κόστος επαναταξινόμησης των οχημάτων όταν, υπάρχει, όταν κάποιος φεύγει από μια χώρα και πάει σε ένα άλλο κράτος μέλος, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει μεγαλύτερο διοικητικό άχθος και γραφειοκρατία. Ε, συμφωνώ το πέρα με τον κύριο Ντεμπάκερ για το χρονοδιάγραμμα, το, το, το χρονικό περιορισμό. Ε, μιλήσαμε για εννέα μήνες όμως, όχι για τρει μήνες. Ε, η πρόταση της Επιτροπής ήταν έξι μήνες. Νομίζω ότι για να διευκολύνουμε τους πολίτες, θα πρέπει να αφήσουμε το μεγαλύτερο ε, δυνατό χρονικό διάστημα, ούτως ώστε όταν κάποιος μετακομίζει, πηγαίνει σε μια άλλη χώρα, πολύ εύκολα μπορεί να δώσει προτεραιότητα σε άλλα ζητήματα. Να αγοράσει ένα σπίτι, ε, μια νέα δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τους αφήσουμε το μεγαλύτερο δυνατό περιθώριο ευελιξίας. και τον απαραίτητο χρόνο για να μπορέσουν και οι πολίτε να ε, χειριστούν αυτό το ζήτημα. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Πέρκερ για την πολύ καλή του δουλειά. Ευχαριστώ, Ρέλα Σέντερ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπίρκεν για όλη αυτή τη δουλειά που έκανε στην γνωμοδότηση σε ένα θέμα που μπορεί να αποτελέσει μια βοήθεια για όσους, όσους ασχολούμαστε με τα θέματα των μεταφορών. Ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τη δυνατότητα διατήρησης της τροπολογίας 31 επειδή ακριβώς λοιπόν ακόμα αναζητάμε την καλύτερη εφαρμογή των προστήμων που είναι διασυνοριακά, κάτι το οποίο όπως ξέρετε ακόμα δεν έχουμε πετύχει αυτό που θέλουμε σε επίπεδο Συμβουλίου. Για να υπάρχει λοιπόν κάποια έτσι αποδοχή είχα καταθέσει μια πρόταση λέγοντας ότι η ταξινόμηση σε μια χώρα σε περιπτώσεις όπου έχουμε εκκρεμότητες ε, πληρωμής ε, προστήμων που δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια να ζητήσουμε, αλλά αν ένα άτομο, το ίδιο άτομο, επιστρέφει στην χώρα όπου έγινε η παράβαση, του ζητάμε με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, που του ζητάμε αναδρομικά την πληρονομή των προστήμων, μήπως ακριβώς λοιπόν το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στην περίπτωση ταξινόμησης των αδειών κυκλοφορία, Δηλαδή να κοιτάξουμε όταν δίνουμε την άδεια κυκλοφορίας αν υπάρχουν ε, προπαρχουσε ε, παραβάσεις και να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ένα παραπάνω εργαλείο πίεσης για την εφαρμογή. Ευχαριστώ. Κ. Κρόμερ. Ο κύριος η Λίχτενμπεργκ δεν είναι εδώ. Εξ ονόματός της θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή ερωτήσεων, κύριε Σκόκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεση. Θεωρούμε ότι η έκθεση αποτελεί ικανή απάντηση, άξια απάντηση στην πρωτοβουλία μας. Παρά τις ε, αντιπροτάσεις, ε, εμείς θα επιμείνουμε στη δική μας πρόταση. Σε ορισμένε περιπτώσεις, κάποιες από τις προτάσεις, ε, ειδικά όσον αφορά το χρονικό διάστημα για την ταξινόμηση και, και λοιπά, τρεις ή εννέα μήνες, υπάρχουν, υπάρχει διάσταση απόψεων, εμείς προτείνουμε τους έξι. Τώρα, όσον αφορά τα σχόλια που ακούσαμε πριν από λίγο, και δει την αναφορά στην οδηγία του 2011, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να απορρίψουμε την ταξινόμηση ακριβώς επειδή υπάρχει μηχανισμός επιβολής της ίσπραξης των προστήμων. Αλλά ε, εκτός από αυτό, ευχαριστώ εν για μια πολύ επικοδομητική προσέγγιση της πρότασής μας. Ευχαριστώ. Πάω σχόλια. Χωρίς μικρόφωνο. Και ο Σπίρκερ χωρίς μικρόφωνο. Εν συντομία για τα δύο αυτά σημεία. Όσον αφορά το εν λόγω χρονικό διάστημα, είχα προτείνει η συμβαστική λύση. Φυσικά, μπορεί ο να βάλει όσο θέλει. Ε, μπορούμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε μήνες από αυτό το χρονικό διάστημα. Κάποιοι είπαν από 3 έω εννέα μήνες. Κάποιοι μένουν μέχρι και 12. Εγώ πιστεύω ότι εντός 6 μηνών είναι απολύτως δυνατόν να καταχωρήσει κανείς, να ταξινομήσει κανείς το όχημά του. Φυσικά υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, το να βρεις ας πούμε, σπίτι, αλλά 6 μήνες είναι υπεραρκετό διάστημα για να γίνει και αυτή η δουλειά. Γι' αυτό και τροποποίησα την πρόταση και μπορώ να συμφωνήσω με την Κομισιόν. 6 μήνες. Κατά δεύτερο λόγο, αιτίες απόρριψης. Εγώ διαφωνώ με την πρόταση που έγινε, διότι θα μπορούσε να συνεπάγεται περαιτέρω καθυστερήσεις, περιττές καθυστερήσεις. Ενώ οι πραγματικέ αιτίε βρίσκονται αλλού. Μόνο και μόνο δηλαδή επειδή η δημόσια διοίκηση ασχολείται με άλλα. Εδώ όμω μιλάμε για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Ο λόγος αυτός λοιπόν του διοικητικού φόρτου της δημόσιας δίκης δεν είναι επαρκής αιτία. Εδώ κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Προσπαθούμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία στο μέγιστο δυνατό βαθμό, κατά τη διαδικασία δηλαδή ταξινομή σε μια άλλη χώρα μέλος. Και αυτό θέλουμε, επαναλαμβάνω, να διευκολύνουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Γι' αυτό ακριβώς πρότεινα οι σκιώδεις να απορρίψουν τη συγκεκριμένη πρόταση. Οπότε θα επιμείνω και εγώ, επί της μου πρόταση, να απορρίψουμε δηλαδή την αντιπρόταση προ όφελο των καταναλωτών. Ευχαριστώ όλου όσου πήραν μέρο στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίρκα. Η ψηφοφορία αύριο το πρωί. Δεν ξέρω πότε θα γίνει η ψηφοφορία στην ΕΜΚΟ, αλλά για μας είναι αύριο. Μετά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, Οπότε ελπίζω ότι θα έχετε επιβιώσει ώστε να έχετε δύναμη να σηκώσετε το χέρι σας και να ψηφίσετε. Αύριο επαναλαμβάνω το πρωί. Πολύ ωραία. Και Καμάλ θα έρθει. Έχει κανείς μια ιδέα πότε θα εμφανιστεί. Εδώ λέει τέσσερις. Έχετε δίκιο. Είναι, δεν είναι ακόμα τέσσερις. Προτείνω να περιμένουμε 10 λεπτά όσο το έρθει και να ξεκινήσουμε. 10 λεπτά λοιπόν διάλειμμα. Uh, uh, Συνάδελφοι, ο κύριος Καμάλ δεν θα έρθει τελικά, όμως η κυρία Φώστερ θα τον αντικαταστήσει. Επομένως, έχουμε πιο όμορφη ύπαρξη μαζί μας σε σχέση με τον κύριο Καμάλ. Αυτό είναι καλό. Το επόμενο σημείο λοιπόν είναι η γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα περιμένω μια στιγμή, γιατί γίνονται κάτι συζητήσει αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δυστυχώ ο συνάδελφο κ. Καμάλη δεν μπορεί να βρίσκεται σήμερα μαζί μα. Ε, για να εξετάσουμε τις τροπολογίε στην Επιτροπή. Όμως θα ήθελα να διαβάσω αυτό που είπε, ότι έχει λάβει υπόψη τα όσα έχουν αναφερθεί και σε πολλέ περιπτώσεις ήταν ε, πολύ σημαντικές και ευχαριστεί τα μέλη της Επιτροπής ε, για τη συμμετοχή του, τη συμβολή τους. Μπορούμε να έχουμε ησυχία παρακαλώ. Ωραία. Ε, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για το κείμενο με τις οποίες συμφωνεί. Ε, για τις πιο αμφιλεγόμενες ε, παραγράφους προσπαθεί να καταλήξει σε συμβιβασμό όπου αυτό είναι δυνατόν ε, και ελπίζει οι συμβιβαστικέ να γίνουν αποδεκτές από την πλειοψηφία των μελών. Ε, εύχεται να μπορούμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς την Επιτροπή Εικόν ότι ο ανοιχτό ανταγωνισμό θα ε, ανοίξει το δρόμο για νέε θέσει εργασία και να αυξήσει την ευημερία σε αυτέ τι ε, δυσμενεί ε, συνθήκε για τους ε, εισηγητές. Θα ήταν καλό να ε, μιλήσουν τώρα, να πάρουν το λόγο για τις συμβιβαστικέ τροπολογίες που έχουν ε, γίνει για να μας ενημερώσουν για τη στάση τους και μετά μπορώ και εγώ να το μεταφέρω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. you, Jackie, for Ευχαριστώ, Τζάκι. Ο κύριος Μπακ. Sorry, I thought Mr. Ja, vielen Κύριος Γκρός, ευχαριστώ πολύ. Σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ο συνάδελφος Λίστα Κανά δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά ε, έθιξε ένα σημείο ότι υπάρχουν πολλοί συμβασμοί και κατά τη γνώμη του, ε, αποτελούν ένα πολύ καλό, ε, έχουμε βρει μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ της, ε, του ανοίγματο αγοράς και διαμόρφωσης μεταφορικού χώρου, χώρου μεταφορών, το οποίο είναι πολύ θετικό, αλλά πρέπει βεβαίω να υποστηρίζεται και από ε, κανονιστικά μέτρα, γιατί η αγορά δεν μπορεί να λύσει και τα δύο αυτά τα προβλήματα. Ε, πρέπει να μπουν λοιπόν κάποιε πιο, κάποιες πιο αποχρώσεις σε ό,τι αφορά τι ε, συνθήκε εργασία, για παράδειγμα και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Έτσι κι αυτό πρέπει να είναι ένα στόχο, ε, η δημιουργία της εργασία και η βελτίωσή του είναι πιο σημαντικό αυτό από το άνοιγμα της αγοράς ως αυτό σκοπό. Μετά, το, το θέμα των ε, κυρώσεων θα πρέπει να συζητηθεί. Θεωρούμε ότι ένας ενιαίος χώρος μεταφορών ε, δεν εξαρτάται μόνο από το άνοιγμα της αγοράς, αλλά και από κοινού και εναρμονισμένους κανόνες ε, και κυρώσεις παντού. Τις κυρώσεις λοιπόν θα πρέπει να, οι κυρώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται και να επιβάλλονται με όμοιο τρόπο σε όλα τα κρατημέλη. Ενώ πολύ συχνά βλέπουμε ότι σε μια χώρα ε, μια παράβαση του κώδικα δικής κυκλοφορίας ε, είναι επισύρει χαμηλότερη ποινή από ό,τι σε κάποια άλλη και η οικονομική πτυχή είναι σημαντική. Πρέπει λοιπόν οι παραβάσεις αυτές ε, να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, Ευχαριστώ, Μπένιεν. Yes, my comments are... Ναι, και εγώ να σχολιάσω μόνο τον Σεβασμό 2 γιατί μόλις λάβαμε μια εκδοχή του. Πριν να τη λάβουμε, ήθελα να πω ότι συμφωνούσα με όλες τις ε, συστάσεις για την ψήφο και τους συμβασμούς. Τώρα όμως πια δεν ισχύει αυτό. Ο συμβασμός 2, η συμβαστική πρόταση 2, καλεί την Κομισιό να ολοκληρώσει την εφαρμογή του ενιαίου συνδρομικού ευρωπαϊκού χώρου και να ανοίξει ο χώρος αυτός στον ανταγωνισμό. Τώρα, η τροπολογία 35, η δικιά μας που βρισκόταν σε αυτό το συμβασμό, ε, δίδει ιδιαίτερη έμφαση στις εσωτερικέ αγορές υδροδρόμων. Όμως η διεθνή αγορά επιβατών και αγαθών, αυτό δηλαδή το οποίο μας αφορά εμάς, ε, δεν λέει κάτι τέτοιο, γιατί οι περιορισμοί μόνο για την ενιαία, για, συγγνώμη, για την εσωτερική αγορά. Τον ζητάμε λοιπόν τώρα εμεί ότι οι τομεί που ήδη ανοιχτοί σε ανταγωνισμό να ανοίξουν σε ανταγωνισμό και αυτοί που δεν ανοιχτοί σε ανταγωνισμό να μην ανοίξουν σε ανταγωνισμό, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε τίποτα. Έχουμε λοιπόν μια συμβαστική πρόταση που δεν έχει πια νόημα, δεν είναι λογική, γιατί στην ουσία καταγράφει και επαναλαμβάνει αυτό που ήδη υπάρχει, την πραγματικότητα δηλαδή. Γι' αυτό ακριβώ στην τροπολογία μα 35 ε, βλέπω ότι αυτή δεν είναι πια τμήμα τη συμβαστική ε, πρόταση και αν παραμένει ο κατάλογο πληροφορία όπω έχει, δηλαδή να λέμε ότι το 35, η 35 μα είναι τμήμα του συμβασμού, ωραία αλλά βλέπω ότι στην τελευταία της ε, εκδοχή αφαιρέθηκε. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ναι, κοιτάξτε. Ο ορισμός της συμβαστικής πρότασης αφορά πάνω από μία ομάδα. Αν έχουμε λοιπόν μία-δύο ομάδες δεν έχουμε μόνο συμβασμό. Η κυρία Τίκα. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι λυπάμαι που δεν είχα καμία συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές και λυπάμαι πραγματικά που δεν ξεκινήσαμε κάποια συζήτηση για αυτό το θέμα. Γιατί νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε καταλήξει σε κάποιους συμβασμούς που θα ήταν αποδεκτοί από όλους και να έχουμε τελικά μια γνωμοδότηση η οποία θα αντανακλά την άποψη της πλειοψηφίας των συναντέλφων της Επιτροπής μας. Πάντως θα ήθελα να πω ότι ως θέμα αρχής οι τροπολογίες και οι συμβαστικές τροπολογίες παρόλο που αφορούν κάποιες τροπολογίες και των σοσιαλιστών αυτές τελικά δεν περιλαμβάνονται στις συμβαστικές προτάσεις. Πιστεύουμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που δεν περιλαμβάνονται στις συμβαστικές προτάσεις θα έπρεπε να ψηφιστούν χωριστά. Και οι συμβαστικές τροπολογίες που λάβαμε δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες σε σχέση με το ποιες πολιτικές ομάδες υποστηρίζουν αυτές τις τροπολογίες. Οπότε, όπως έλεγε και ο πρόεδρος πριν από λίγο, ε, εδώ έχουμε συμβαστικές τροπολογίες, αλλά θα πρέπει να ψηφίσουμε τον κατάλογο με τις τροπολογίες οι οποίες είχαν κατατεθεί από τους δικούς μας συναδέλφους. Έχουμε εδώ εξάλλου και κάποιες ε, τεχνικές αναφορές σε σχέση με την γνωμοδότηση και να πω ενδεικτικά ότι ως θέμα αρχής δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την απελευθέρωση τη στιγμή που έχουμε και την εμπλοκή κοινωνικών θεμάτων και παραγόντων. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν δίκαιο ανταγωνισμό και αυτό ο δίκαιο ανταγωνισμό να αφορά και τα κοινωνικά θέματα, σαν να διασφαλίζονται αυτά. Δεν είμαστε λοιπόν υπέρ τη απελευθέρωση σε αυτού του τομεί. Γιατί πιστεύουμε ότι θα έπρεπε εδώ να λάβουμε υπόψη μα και άλλα κόστη που αφορούν συνθήκες κοινωνικές, συνθήκες που αφορούν την απασχόληση γενικότερα κλπ. κλπ. Εγώ ίδια ε, κατέθεσα τροπολογίες σε σχέση με τον τομέα των μεταφορών και μάλιστα ζητήσαμε από την Κομισιόν να δει κατά πόσο υπάρχουν συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ιδιαίτερα ε, όσον αφορά τους μεταφορείς χαμηλού κόστους. Να πω πάντως ότι είμαστε υπέρ των περιφερειακών και θεωρούμε ότι αυτοί οι αερολιμένες περιφερειακοί θα έπρεπε οπωσδήποτε να περιληφθούν στην πολιτική που αφορά την εσωτερική αγορά της κάθε χώρας. Επίσης είχαμε και κάποιες ε, προτάσεις όσον αφορά την απελευθέρωση των οδικών μεταφορών και να πω ότι επ' αυτού συμφωνούμε με τις τροπολογίες οι οποίες λένε ότι αυτή η απελευθέρωση θα πρέπει να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου τηρούνται συγκεκριμένοι κοινωνικοί κανόνες και προϋποθέσεις. Και μόνο τότε θα έπρεπε να προχωρήσουμε. Θα σταματήσω εδώ πάντως. Λυπάμαι για το γεγονός ότι θα γίνει αύριο η ψηφοφορία, αλλά εμείς ακόμα σήμερα δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο κατάλογο ψηφοφορίας. Θα ψηφίσω αύριο βεβαίως, αλλά λυπάμαι γιατί οι συμβαστικές προτάσεις δεν ξέρω πόσες πολιτικές ομάδες τις ε, υποστηρίζουν. Ο εισηγητής θεωρεί ότι κάποια τμήματα εδώ δεν καλύπτονται. Και αυτά τα τμήματα που δεν καλύπτονται και έχουμε τροπολογήσει, αυτά θα πρέπει να ψηφιστούν ε, χωριστά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, συνήθω πριν από μια ψηφορία συγχαίρουμε τον εισηγητή. Αδύνατον όμω. Ε, προκειμένου δεν τον γνωρίζω, δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν ε, ενημερωθήκαμε. Δεν μας είπε ποτέ για την υπέρ κατά κάποιας τροπολογίας. Πραγματικά ε, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναζήσει. Και δεν είναι καν εδώ σήμερα που συζητούμε την έκθεσή του. Ε, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν είναι συνεργασία. Καταλαβαίνετε, ε, μετά από 7 χρόνια ζω κάτι το οποίο βρίσκω εξοργιστικό. Έχουμε εδώ να συζητήσουμε μεταξύ άλλων τον αθέμητο ανταγωνισμό στον τομέα των μεταφορών. Ο Σίγητης συνέχισε να δρά με παροπίδες Μάλιστα ο Γιώχανες Λούντβιχ από την Τσεντεού, του συντηρητικού στην ε, Γερμανία, είπε ότι είναι σαν να μην ισχύει στον τομέα των μεταφορών ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Να μην υπάρχει εσωτερική αγορά. Όλα αυτά φέρονται σαν μια σταλινιστικού τύπου δολοπλοκία. Δείτε ας πούμε, τις ε, θέσεις του όσον αφορά τα αεροδρόμια, τα οποία πετούν δύο πτήσεις την εβδομάδα. Και κάποιοι λένε ότι δεν μπορούμε να τα κλείσουμε γιατί επενδύσαμε και τώρα πρέπει να επενδύσουμε ακόμη περισσότερα, αν χρειάζεται να τα κλείσουμε. Δείτε το Στρασβούργο, τις συνδυοδρομικές μεταφορές, δείτε την EasyJet, η οποία μας λέει ότι έβγαλε 300 εκατομμύρια, ενώ στην πραγματικότητα έχουν χάσει, έχουν ζημίες 500 εκατομμυρίων. Τα 807 εκατομμύρια διαφορά είναι επιδοτήσεις. Το, οι ίδιοι το λένε αυτό. Λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι πρέπει τα αεροδρόμια να τα αξιοποιούμε καλύτερα και αυτό δεν έχει σχέση με ανταγωνισμό. Αν και στην πραγματικότητα πρόκειται για στρέβλωση του ανταγωνισμού. Είναι μια κεντρικά σχεδιαζόμενη οικονομία. Εκεί έχουμε γυρίσει. Αφήστε που καταστρέφουμε και το περιβάλλον. Αν θέλουμε επενδύσει, να τι κάνουμε. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε κάποια υγιή επένδυση μα λένε δεν έχουμε χρήματα. Ύστερα δεν έχουμε καν διασυνοριακές σιδηροδρομικές μεταφορές. το EFA δεν ε, λειτουργεί. Αν θέλουμε οι χώρε μα να αναπτύσσονται αντίστοιχα λίγο πολύ με τον ίδιο ρυθμό, χρειαζόμαστε περισσότερε διασυνοριακέ μεταφορέ. Και εκεί, για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε απελευθέρωση του συστήματο. Εγώ είμαι Ευρωπαίο, σκέφτομαι ευρωπαϊκά. Δεν μπορούμε λοιπόν να δυσκολεύουμε, παραλαμβάνω, τι διασυνοριακέ μεταφορέ και συνδέσει. Τώρα, όσον αφορά την διευκόλυνση του ανταγωνισμού. Σε μία από τι τροπολογίε που αναφέρεται, και στην 10 συγκεκριμένα, η οποία νομίζω έχει απορριφθεί. Δεν ξέρω μάλιστα γιατί απορρίφθηκε. Γιατί είναι σαφέ το εξή. Εάν θέλουμε, επαναλαμβάνω, να διευκολύνουμε την περιβαλλοντικά φιλική αεροπλοεία και τις αντίστοιχες συνδυοδομικές μεταφορές, μας λένε κάποιοι ότι πρέπει να πάρουμε αυτοκίνητα από τους δρόμους για να ευνοήσουμε τους άλλους δύο τομείς. Εδώ η ΣΥΙΤΙΣ δεν μας λέει τίποτα. Ίσως καλύτερα γιατί δεν έχει τίποτα χρήσιμο να πει. Συγγνώμη που είμαι αυστηρός και επικριτικός, αλλά αυτή είναι η κατάσταση, πολύ φοβούμαι. Πρόεδρε, ο συναδελφός μας, ο κύριος Γκρός, είπε αυτά που όφιλε να πει. Εγώ δεν θα επιμείνω ότι θα σχολιάσω τις συμβαστικές τροπολογίες. Να πω όμω δύο λόγια, απλώς για το πακέτο ότι δέσμη μέτρων που αφορούν τα αεροδρόμια και για τον φόρο για το τροχαίο υλικό στην Γαλλία. Στη Γαλλία το σύστημα λειτουργεί μάλλον ικανοποιητικά. Δεν είναι 100% ικανοποιητικό, τέλειο, αλλά εγώ είμαι ικανοποιημένο. Πέραν αυτού όμως, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι εξέφρασα την ικανοποίησή μου για την επιστολή από τον πρόεδρό μας προ τον αρμόδιο επίτροπο, ε, με την οποία ζητούσε να πάρει θέση επιτέλου η Επιτροπή επί του θέματος. Δεύτερον, σχετικά με αυτό το οποίο είπε ο Ματιέ, κυρώσει σε περιπτώσει σοβαρών παραβάσεων των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των μεταφορών. Ο Αυστριακός συνάδελφος το 2010 εκπώνησε σχετική έκθεση όπου διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρκετά αυστηρή. Με άλλα λόγια, η ενερμόνιση δεν έχει ολοκληρωθεί προκειμένου και κάποια κατημέλη όντως δεν τηρούν, δεν ε, σέβονται τους εφαρμοστέους κανόνες. Σε ορισμένε χώρε υπάρχουν κυρώσει, ολόκληρο κατάλογος κυρώσεων, πολύ διαφορετικέ ε, όμως από αυτές σε άλλε χώρε. Συνεπώς, χρειαζόμαστε περισσότερη εναρμόνιση στον τομέα. Ε, σε ορισμένε ε, χώρες ε, οι κυρώσει δεν λειτουργούν προοδευτικά, σε ναι. Μετά η φύση της κύρωση είναι χρηματική αλλού διαφορετική. Χρειάζεται λοιπόν περαιτέρω παραλαμβάνω εναρμόνιση όσον αφορά τι κυρώσει. Υφίστανται φυσικά κάποιε διατάξεις, οι εφαρμόζεται με πολύ διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα. Και αυτό αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ο Ματιού μίλησε και για, την τέταρτη δέσμη μέτρων για του σιδηροδρόμου. Εδώ θεωρώ ότι χρειάζεται προσοχή. Φοβούμαι ότι ανοίγουμε έτσι το κουρί της Πανδώρας. Εφτά χρόνια κάναμε να καταλήξουμε στη συμφωνία προκειμένου. Και το λέω διότι γενικώ το άνοιγμα τη αγορά. Είναι καλή ιδέα, ακούγεται καλή ιδέα, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και το κοινωνικό κομμάτι. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γρηγοροβίτ από την Επιτροπή. Πριν ξεκινήσετε, κύριε Γρηγοροβίτ, με προβληματίζει το γεγονό ότι δεν υπήρξε συνεδρίαση των σκιωδών και δεν υπήρξε συνάντηση ε, για την εξέβρεση συμβιβασμών. Επομένως, θα πρότεινα να αναβληθεί, αλλά θέλω πρώτα να ακούσω τον κύριο Γκρικόροβιτς. Ήθελα να σας τα πω αυτά πριν πάρετε το λόγο. Έχετε το λόγο, απλώς να έχετε κατά νου αυτά που σας είπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω να απαντήσω σε δύο ζητήματα που αναφέρθηκαν ε, στην προηγούμενη συνεδρίαση τον Νοεμβρίο, στις 6 νομίζω. Το ένα αφορούσε ε, τη συμφωνία με τις αεροπορικές εταιρείε και τους κανόνες ανταγωνισμού και το δεύτερο για το e-fair, για το συντροδρομικό δίκτυο. Ξεκινήσω με το πρώτο. Ε, νομίζω ότι η απάντηση του κύριο Κίνης έχει ήδη αποσταλεί, αλλά θα την ξαναδιαβάσω. Στις 6 Νοεμβρίου λοιπόν το ζήτημα αυτό γιατί με τη μείωση των αγωνισμού στις αεροπορικές εταιρείες ε, ε, ε Η Επιτροπή εξετάζει δύο περιπτώσεις για να δει αν οι συμφωνίες αυτές ε, ευθυγραμμίζονται και συνάδουν με τη, με το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είχαμε συμφωνία Λουφτχάνσα ε, και ε, τουρκικών αερογραμμών, αλλά και των Brussels με την πορτογαλική εταιρεία. Οι κοινέ πτήσει λοιπόν είναι μια κοινή πρακτική βεβαίω στη βιομηχανία αυτή. Συνήθω όμω γίνεται από μία αερογραμμή, αλλά ε, η εμπορία γίνεται από άλλη. Ε, οι κοινέ πτήσει μπορούν να έχουν σημαντικά ωφέλη για του ε, επιβάτε. Κάποιε μορφέ όμω μπορούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό. Οι συνεχιζόμενες λοιπόν έρευνες αφορούν μια μορφή τέτοια συμφωνίας κοινών πτήσεων όπου και οι δύο έχουν αναλάβει τις πτήσεις και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των ε, θέσεων που μπορεί να πουλήσει ε, η μία εταιρεία στις πτήσεις της άλλης. Σε τέτοιες ε, μορφές συμφωνίας μπορεί να υπάρξει μείωση του ανταγωνισμού σε αυτές τις ε, ε, συνδέσεις με αύξηση των τιμών και μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές. Εάν αποδειχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, τότε η Επιτροπή μέσω της έρευνάς της θα έχει ως στόχο να, να δώσει σωστές κατευθυντήριες γραμμές και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για το τι ε, ακριβώς περιλαμβάνουν οι κανόνες ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκής οι αεροπορικές γραμμές θα πρέπει να ε, εξετάσουν αν θα πρέπει οι συμφωνίες τους να ε, τροποποιηθούν ακόμα και αν ε, δεν συμπεριλαμβάνονται σε έρευνα της Επιτροπής. Το δεύτερο για το e-fair υπήρξαν διαβουλεύσεις με την Γενική Διεύθυνση MOVE. Οι, επιτρο... οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν την επιβολή ενιαίου ε, φόρου στη Γαλλία για οτιδήποτε χρησιμοποιείται στο συνδρομικό δίκτυο της Γαλλίας θεωρεί η Επιτροπή ότι αυτός ο φόρος στη Γαλλία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αγορά για τις υπηρεσίες επιβατών γιατί αυτό μπορεί να να εμποδίζει τους ε, εξωτερικούς εμπορευομένους να παρέχουν υπηρεσίες στη Γαλλία ή μέσω της Γαλλίας. Και η Επιτροπή θα κάνει τα απαραίτητα βήματα για να ε, διασφαλίσει ότι ε, ακολουθούνται οι κανόνες που εγγράφονται στις συνθήκες λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάικλ, το θεωρώ θετικό που η Επιτροπή βλέπει ότι υπάρχει απειλή για, την, για τον ανταγωνισμό, αλλά πάνε δύο χρόνια που περιμένουμε για μια απόφαση. Περιμένουμε και θα είναι πολύ αργά αν καθυστερήσουμε κι άλλο. Γιατί η Επιτροπή λοιπόν περίμενε μέχρι τώρα. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση εδώ και δύο χρόνια. Και τώρα ακούμε μια δήλωση. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς κάνει εδώ η Επιτροπή. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Μάικ, μιλάς για το φόρο για τους γαλλικούς σιδηρόδρομους. Κομισιόν θέλετε να απαντήσετε μήπως. Τώρα θα καταγράψω το έτοιμά σας και θα σας απαντήσουμε στη συνέχεια. Μπορεί να, γράφουμε, μπορεί να απευθυνόμαστε στο λάθο άνθρωπο, λέει ο πρόεδρος, αλλά τέλο πάντων. Αν σκοπεύουμε να ψηφίσουμε αύριο, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους κοιόδης, τις συναντήσεις τους, τις μη συναντήσεις τους, τους συμβαστικούς, ε, συμβαστικές τροπολογίες, προτάσεις κτλ. κτλ. Μου είπαν ότι η Επιτροπή θα ψηφίσει το Φλεβάρι. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία, αν συμφωνείτε, να αναβάλουμε την ψηφοφορία αυτή για τις 26 του Γενάρη και σας προτείνω αυτό ακριβώς να κάνουμε. Συμφωνείτε λοιπόν να κάνουμε μια μετατόπιση και να στείλουμε μήνυμα στον εισηγητή να συναντηθεί με τους σκιώδεις έτσι, μετά τα Χριστούγεννα και να προχωρήσουμε έτσι. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, καλή πρόταση. Ο Σαΐτ είναι άρρωστος. Και αυτό ακριβώ το λόγο απουσιάζει σήμερα. Και να πω ότι μου προκαλεί έκπληξη ότι ο κ. Κράμερ που, ήταν, που είναι χρόνια μέλος εδώ λέει ότι απουσιάζει ο Αυτό δεν είναι σωστό. Ο κ. Καμάλ ξαναλέω είναι άρρωστος. Αρρώστησε σήμερα. Του έστειλα μήνυμα και θα στείλει κάποιες πληροφορίες στο γραφείο του εδώ το θέμα αφορά βεβαίως τους συμβαστικούς, ε, τους συμβασμούς, συμβαστικές προτάσεις. Βλέπω ε, και καταγράφω αυτό που είπε ο Πρόεδρος ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Αποδέχομαι λοιπόν την πρόταση του Προέδρου να αναβάλουμε ψηφοφορία για τον Γενάρη. Και είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Καμάλ θα έρθει τότε. Ζητά λοιπόν συγγνώμη για την απουσία του και αν επιτρέπετε να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση με τις κοινέ πτήσει. Δεν ξέρω αν βρίσκομαι σε άλλο πλανήτη, αλλά το code sharing, κοινέ πτήσει υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια και βάλε. Δεν ξέρω λοιπόν τι λέει ο καλός συνάδελφος από την Κομισιόν. Όταν υπάρχουν κοινέ πτήσει μεταξύ διαφόρων εταιριών, ξέρουμε ότι αυτή είναι συνήθις πρακτική. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν εδώ στην ε, γνωμοδότηση. Μου προκαλούν έκπληξη τέλο πάντων όλε αυτέ οι λεπτομέρειε, ενώ εμεί θα πρέπει να κάνουμε δράσει και θα πρέπει να προωθήσουμε ακριβώ τι κοινέ πτήσει στα περιφερειακά αεροδρόμια ώστε να επιβιώσουν και επιχειρήσει και τα αεροδρόμια. Αλλά τέλο πάντων, θα ξανασυζητήσουμε με την Κομισιόν για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πρόταση πάντως, για την πρόταση πάντω, Πρόεδρε, και νομίζω ότι είναι καλύτερη, καλύτερη η ψηφοφορία τον Γενάρη. Ευχαριστώ. Μάικλ. Ναι, εγώ δεν παραπονιόμαι για το γεγονό ότι απουσιάζει σήμερα. Εντάξει, σήμερα. Αλλά αυτό έχει ξαναγίνει κάμποσε φορέ στο παρελθόν, να αποσιάζουν λόγω ασθένεια. Εγώ είπα ότι δεν υπήρχε συνάντηση, δεν είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε στους ε, σκιώδεις. Αυτή την ευκαιρία χάσαμε. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπω στα 7 χρόνια παρουσίας εδώ στην Επιτροπή. Αυτό είπα στα σχολεία μου. Εντάξει, λέει ο πρόεδρο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα αναβάλουμε την ψηφορία ώστε να είναι παρόν και ο εισηγητή, να έχει συναντήσει ενδιάμεσα και του ε, σκιώδει και το αναβάλουμε λοιπόν για τι 26 του Γενάρη. 27 του Γενάρη. Ωραία. Θα σας ζητήσω τώρα να φύγετε από την αίθουσα όσοι δεν είσαστε συντονιστές και όσοι δεν είσαστε συντονιστές, τα μέλη της Επιτροπής, να φέρετε την κάρτα ψηφοφορία σας αύριο. Γιατί αν δεν έχετε την κάρτα δεν θα μπορείτε να ψηφίσετε. Έτσι να είναι αυτό ξεκάθαρο. Δεν θέλω να βλέπω χεράκια να σηκώνονται και να λένε και εγώ και εγώ. Ωραία άδειας και θα συνδράσουν σε λίγο συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ.